Γεια σας συνάδελφοι, ε, καλό απόγευμα, συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να προβώ σε κάποια ανακοίνωση όσον αφορά τα χθεσινά πρακτικά.